που είναι δημοσιογράφος, πολιτικός και πρόεδρος της Ένωσης των ε, Γυναικών Δημοσιογράφων, αδέσμευτων γυναικών δημοσιογράφων, καθώς και συντονιστής ε, της εξέγερσης ε, των νέων στην Ιεμένη. Είναι μία από τις τρεις γυναίκες που θα λάβουν Εντό ολίγου ε, το Νομπέλ ε, για τον μη ε, το Νομπέλ Ειρήνη, συγγνώμη, για τον μη βίαιο αγώνα για την ασφάλεια των γυναικών και τα δικαιώματα των γυναικών. Την περασμένη εβδομάδα πήγα στην Τουρκία για την επίσημη επίσκεψη ε, προσφώνησα το κοινοβούλιο, συναντήθηκα με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, μίλησα με τον Πατριάρχη Βαρθολομέ για την κατάσταση των χριστιανών στην τουρκία θέλουμε να αναζωογονήσουμε